συνθήκες πλαίσιο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 Τώρα περνούμε σε προσώπους των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους ε, του ΕΛΚ πρώτη θα λάβει το λόγο η κυρία Σοφία Ριμπέιρο.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 Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει ο κύριο Νικολά Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα ζώα είναι ε, ε, όντα που αισθάνονται.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 ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκε μεταφοράς ε, των ζώων ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ε, συντομεύοντας τη διάρκεια των μεταφορών στις 8 ώρες από την κτηνοτροφική μονάδα στο σφαγείο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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθημερινά, εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται σε φορτηγά αεροπλάνα και καράβια στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η Ευρώπη είναι περίπου στο 100% τη συμμόρφωση με του ευρωπαϊκού κανόνε τη νομοθεσία για τη μεταφορά των ζώων. Ε, το επανέλαβε και σήμερα το πρωί. Είναι απολύτω αναλυθέ αυτό. Είναι ψεύδο.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 πρόσφατα το καλοκαίρι πήγα και σε μια αποστολή στην Κροατία και τα είδα και με τα μάτια μου. Ε, τα φόρτηγα δεν ήταν κατάλληλα. Τα ζώα βρίσκονταν ε, σε συνθήκες ε, φοβερής ζέστης. Πολλές φορές ήταν πληγωμένα και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 Πώ ε, θα ποτιστούν ή θα πιούν Επίση, Επίσης, ότι οι ζώα που μεταφέρονται προ την Αφρική ε, βρίσκονται σε μια κόλαση μετά από μια, ένα φρικαλαίο ταξίδι. Πότε θα αρχίσετε να παίρνετε στα σοβαρά τι ανησυχίε εκατομμυρίων πολιτών ε, και του Ευρωκοινοβουλίου. Πρέπει να πάψουν αυτέ οι φρικαλές συνθήκε μεταφορά που επικρατούν σήμερα. δεν έχει γίνει ακόμα σήμερα, αλλά κάτι να γίνει για να πάψουν αυτέ οι πρακτικέ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Πρασίνων, το λόγο έχει ο κύριος Τόμας Βάιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.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 τους ε, συναδέλφους του ΕΛΚΑ που έχουν καρδιά ακόμη και ελπίζουμε να μας υποστηρίξουν. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της FDD, ο κύριος Μάρκο Τσούλο. Καλημέρα, Πρόεδρε.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 Έχουμε τεράστιο αριθμό παραβιάσεων. Δεν γίνονται σεβαστέ οι διατάξει. Καταχρηστική μεταφορά, ακατάλληλο ε, εξοπλισμό, ε, μη αρκετό πότισμα των ζώων, άθλιε συνθήκε, ε, αφιδατωμένα, χωμένα, αποδυναμωμένα φτάνουν τα ζώα, μερικέ φορέ ακροτηριασμένα, εξουθενωμένα, άθλιε καταστάσει. Δεν, δεν, δεν πρέπει να συνεχιστούν. Θα πρέπει να γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι και πιο αυστηρέ κυρώσει για συμμόρφωση με τον κανονισμό. Τούτου η καλύτερη λύση θα ήταν να αποφύγουμε τη μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις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 Μόνο ε, εντό τη ε, κτηνοτροφική μονάδα μεταφέρονται τα ζώα από τον κτηνοτρόφο. Δεν είναι οι κτηνοτρόφοι αρμόδιοι για τη μεταφορά. Εμεί είμαστε υπέρ των ζώων και τα προστατεύουμε. Πρώτα απ' όλα όμω προστατεύουμε του κτηνοτρόφου που τα εκτρέφουν. Και επίση ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ρεαλιστικέ, εφικτέ διατάξει για να διευκολύνουμε τη μεταφορά των ζωντανών ζώων εντό τη Ευρώπη σε κανονικέ συνθήκε. Ευχαριστώ κύριο Στέφανα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Με του κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005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 Μα κοροϊδεύουν κύριε Επίτροπε, πολύ απλά διότι η οδύνη των ζώων δεν του νοιάζει, δεν του ενδιαφέρει, δεν βαρύνει καθόλου απέναντι στο κέρδος της γεωργοδιατροφική βιομηχανία. Αυτό είναι το σκάνδαλο λοιπόν. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, διότι αν δεν ενδιαφέρει το κοινοβούλιο αυτό ή του ηθήνοντε, ενδιαφέρει του πολίτε, τις ΜΚΟ, του δημοσιογράφου. και ε, θα ε, διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με την αδράνεια αυτή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 η οποία έχει οδηγήσει στη σύνταξη αυτής της εξισορροπημένης έκθεσης με λογικές προτάσεις. Η μεταφορά των ζώων των ζώων είναι ένα θέμα που έχει αρνητικέ συνέπειες για όλη την, παραγωγή, την αλυσίδα παραγωγής κρέατος στην Ευρώπη. Συχνά εκτινοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα. Ανησυχούμε λόγω της τρέβλωσης ανταγωνισμού που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Γνωρίζουμε όμως ότι εκεί πρέπει να ε, εντοπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα, το κόστος παραγωγής που έχει να κάνει με την εκτροφή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 Θα υποστηρίξουμε τις εναλλακτικέ της σφαγής των ζώων σε τοπικό επίπεδο για να δοθεί και μεγαλύτερη ενίσχυση στην τοπική κτηνοτροφία, διότι είναι δεν είναι κτηνοτρόφοι υπεύθυνοι, αλλά εμείς, για την ταλαιπωρία των ζώων. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δέκα χρόνια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 των θάνατων εκατομμυρίων ζώων το χρόνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Herbert Dorfman.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 προβλήματα υπάρχουν και τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης ε, υπάρχει και μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, την προσυπογράφουν πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες γιατί δεν συμφωνούν με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο να διερωτηθούμε τι θα κάνουμε συνολικά με αυτή την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, των πολιτών. Θα πρέπει να δούμε επίσης πού δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα και πώς μπορούμε να έχουμε μια τοπική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 Ευχαριστώ. Κατοντάδες χιλιάδες, ε, μάλλον χιλιάδες ε, ε, χιλιόμετρα μεταφέρονται χωρίς αερισμό, χωρίς πότεσμα, τάισμα, με στρες, με φόβο. Αυτό πραγματικά το πεπρωμένο χιλιάδων ζώων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 η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ. Είμαι πραγματικά αγανακτισμένη, εξοργισμένη. Εκατομμύρια ζώα κάθε χρόνο ε, μεταφέρονται σε λεϊνές συνθήκες μεταφοράς. Ε, ε είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης, ε, αντικείμενα κακής μεταχείρισης, απαράδεκτο. Και τα ζώα, όπως και οι άνθρωποι, έχουν δικαίωμα στην καλή μεταχείριση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 μην μας λέτε λοιπόν ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είστε αρμόδιος επίτροπος και για την ε, ευημερία των ζώων και ο αρμόδιος επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει δράση. Επίσης πολλές φορές έχουμε λαθρεμπόριο ε, κατοικιδίων, σκυλών και γάτων από τη Ζεχία προς την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό πέρασε παρατηρητό. Κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προστασία των ζώων κατά την μεταφορά εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης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 Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλόρεν Μπαρτσελές έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε χρόνο πάνω από 400 δισεκατομμύρια 400 δισεκατομμύρια ζώα μεταφέρονται και μερικέ φορέ σε μεγάλε αποστάσει χωρί τροφή, χωρί νερό και ακραίε θερμοκρασίες, σε καύσωνα. Αυτή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 πρέπει να δίνουμε προτίμηση στη μεταφορά σφαγείων ή κρέατος και όχι ζώων των ζώων. Σε περίπτωση όμω που είναι απαραίτητη μεταφορά ζώων των ζώων θα πρέπει να εφαρμόζουμε του αυστηρού κανόνε και τι προδιαγραφέ που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση θα πρέπει να ενισχύσουμε την εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών και αυστηρών κανόνων με τη διενέργεια ελέγχων. Είμαι κατά τη υιοθέτηση νέων κανόνων εφόσον έχουμε αποτύχει να εφαρμόσουμε την υπάρχουσα, την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι ισχύοντε κανόνε είναι αρκετά αυστηροί, αλλά δεν εφαρμόζονται επαρκώ. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τον αριθμό των ελέγχων και επιθεωρήσεων στα σύνορα και να επιβάλλουμε κυρώσει στου παραβάτε, σε όσου δεν τηρούν κατάλληλε συνθήκε μεταφορά.